Καλησπέρα, συνάδελφοι. Συνεχίζουμε. Τη συνεδρία στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο. Καλωσορίζω εδώ τον Υπουργό εκ μέρους της Βελγικής Προεδρίας. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση της κυρίας Βίνκερ Φλούτσε σχετικά με άτομα με αναπηρία και τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Κύριε Υπουργέ, όταν είσαστε έτοιμος, παρακαλώ να απαντήσετε. Madame la Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο δίνει μεγάλη σημασία στην αύξηση δυνατοτήτων απασχόλησης και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία μεταξύ άλλων θέλουμε να συμμετέχουν στην αγορά εργασία. Η στρατηγική 2020 που ενέκρινε στις 17 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο ε, δείχνει ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία θέλη, με μέτρα να φροντίσει για την καλύτερη συμμετοχή στην κοινωνία των ατόμων αυτών. Η στρατηγική 2020 λοιπόν κάνει μνήα των ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας, που έχει επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Και εδώ προσθέτω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ετοιμάσει τα προγράμματα για την καταπολέμηση των διακρίσεων, μεταξύ άλλων και για τα άτομα με αναπηρία. Τα κράτη-μέλη δηλαδή θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν μέτρα που να ανταποκρίνονται στις διατερότητες των ε, ατόμων ε, που έχουν μια ιδιαιτερότητα μεταξύ άλλων και των ατόμων με αναπηρία. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να δράσουν τώρα προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τις προτεραιότητες αυτές στο επίπεδό τους. Οι κοινέ πολιτικές πρέπει να στηρίξουν τη στρατηγική αυτή. Έτσι θα υπάρξει καλύτερη συμμετοχή στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρία, κάτι το οποίο αναφέρεται και στο ψήφισμα που έχουμε για ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για θέματα αναπηρίας που ανέκρινε τον Ιούνιο το Συμβούλιο. Εκεί καλεί τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβουν και τα θέματα ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και να φροντίσουν να αξιολογήσουν το δυναμικό που είναι τα άτομα με αναπηρία και να φροντίσουν για την κατάρτισή τους ώστε να έχουν πιο εύκολα πρόσβαση στην απασχόληση. Επίσης, το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει για την επόμενη δεκαετία και σε συνεργασία με τα άτομα με αναπηρία και τις οργανώσεις που τα εκπροσωπούν μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική υπέρ των ατόμων με αναπηρία που να βασίζεται μεταξύ άλλων στην ε, στρατηγική Ευρώπη 2020. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ, κυρία Μπλίνκριβούτσε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας. Όμως, εξακολουθώ να λέω ότι έχουμε 65 και πλέον εκατομμύρια ανάπηρα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η φωνή τους δεν ακούγεται. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να επιταχύνετε την εφαρμογή της οδηγίας για μέτρα κατά των διακρίσεων από όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορέσουν να ζήσουν σαν όλους τους υπόλοιπους πολίτες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Υπουργός. Κοιτάξτε, η ομάδα εργασία του Συμβουλίου για τα κοινωνικά ζητήματα εξακολουθεί να εξετάζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια νέα οδηγία που θα συμπεριλαμβάνει την αρχή τη ίση μεταχείριση των ατόμων ανεξάρτητα με τη θρησκεία, ε, τι αναπηρίε ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Η έγκριση τη οδηγία αυτή απαιτεί ομοφωνία των ε, χωρών μελών. Πολλές προεδρίες έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες για την πρωτοβουλία αυτή. Σε αυτό το στάδιο η Προεδρία δεν μπορεί να σας πει πόσο θα κρατήσουν οι διαπραγματεύσεις και πότε θα έχουμε αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ευχαριστούμε πολύ, Λε Πρόεδρος. Τώρα έχω δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις ακόμα. Θα τις ακούσουμε με τη σειρά και μετά ο υπουργό θα απαντήσει και στις δύο. Η πρώτη είναι από τον κύριο Ζέμκα. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία που μας δώσατε, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που η πληροφορία αυτή ήταν πάρα πολύ γενική. Εσείς ε, αναφέρατε σωστά πράγματα. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Έχετε κάποια πρόβλεψη για επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Γιατί αν δεν υπάρξουν επιπρόσθετα κονδύλια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε καθορίσει για να αντιμετωπιστούν οι νομοθετικές διατάξεις σε σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών, ε, κυρίως των ε, επιβατών αυτοκινήτων. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Για την χρηματοδότηση θα γίνει μια γενική συζήτηση προφανώς, δημοσιονομικού χαρακτήρα, για τον τρόπο με τον οποίο ο ερχόμενος προπολογισμό, οι ερχόμενοι μάλλον προπολογισμοί θα συμπεριλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες εμβληματικές και κάποιες από τους στόχους που θα τεθούν στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Θα δούμε κατά πόσον σε αυτήν την ε, νέα στρατηγική θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στόχους και για τα άτομα με αναπηρίες. Θα δούμε πώς οι δημοσιονομικοί πόροι μπορούν να ακολουθήσουν και αυτήν την νέα πολιτική προτεραιότητα. Ως προς την εξέλιξη της νομοθεσίας, θα πρέπει να δούμε ξεκάθαρα και πολύ προσεκτικά ποιο είναι ο ρόλο που μπορεί η Επιτροπή να διαδραματίσει σε σχέση με την υπάρχουσα νομοθεσία και βάσει των αρμοδιοτήτων που τη αποδίδονται από τι συνθήκε. Το Συμβούλιο θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προστασία των ατόμων με αναπηρίε. Εδώ και δέκα χρόνια επί παραδείγματι, έχει υιοθετήσει μια οδηγία το Συμβούλιο που απαγορεύει τη κριτική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίε, ιδίω στον χώρο τη εργασία, την απασχόληση. Οπότε προφανώ θα συνεχίσουμε να ε, αναλαμβάνουμε δράση στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα βάσει τη ημερήσια διάταξη από την Αντιπρόεδρο κυρία Κράτσαρ. Δημοσιονομική προσαρμογή και ιδιωτικό χρέο είναι το θέμα. Υπουργέ, όταν είστε έτοιμος. Σε αυτή τη φάση διαδικασίε μακροοικονομικής και δημοσιονομικής επαγρύπνησης βάσει του άρθρου 121 και 126 της Συνθήκης είναι ακρογωνιαίο λήθο του συντονισμού των πολιτικών μας σε οικονομικό επίπεδο. Κατά τη συνάντηση του Μαρτίου 2010, το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δημιούργησα μια ομάδα εργασία με την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με αντιπροσώπου από όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ανέλαβε η ομάδα αυτή να μελετήσει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτεθούν οι στόχοι και να μπορεί να αντιμετωπίζεται καλύτερα η κάθε κρίση που συμβαίνει με δημοσιονομικούς πόρους και προκειμένου να ενισχυθεί και το νομοθετικό πλαίσιο. Η ομάδα εργασία υπέβαλε μια έκθεση ενδιάμεση στο Συμβούλιο του Ιουνίου και στην έκθεσή τη υπογραμμίζει η ομάδα εργασία ότι οι διαδικασίε δημοσιονομική επαγρύπνηση πρέπει να ενισχυθούν ιδίω αποδίδοντας μεγαλύτερη προσοχή στο επίπεδο και την εξέλιξη του χρέους καθώς και την ε, βιωσιμότητά του στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, η ομάδα εργασία εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να εγκριθούν διαδικασίε επαγρύπνηση μακροοικονομική, πιο αποτελεσματικέ, ώστε να εντοπιστούν ε, οι ελλείψει ισορροπία μακροοικονομική σε πρώιμα στάδια και να προληφθούν οι δυσμενείς τους συνέπειες και ο δυσμενείς τους αντίκτυπο Επίσης να οριστούν σαφεί δείκτε γιατί προφανώς το ιδιωτικό χρέος μπορεί να δειχθεί σημαντικός παράγων για όλα αυτά. Στις 6 ε, ε, Ιουνίου και 17 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τους γενικούς αυτούς προσανατολισμούς και η ομάδα εργασία θα υποβάλει την τελική της έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου βάσει των πορισμάτων των εργασιών της προκειμένου να περάσουμε στην έγκριση ενός νέου νομοθετικού κειμένου της Ένωσης ή να διορθώσουμε τα υπάρχοντα νομοθετικά κείμενα. Και Βεβαίω, η, Προεδρία, η Προεδρία θα δώσει ε, προτεραιότητα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία ληφθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε, κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την ε, ε, προσπάθεια απάντηση στην ερώτησή μου, αλλά δυστυχώ δεν κατάλαβα κάτι το οποίο αναφέρεται σε αυτό που ρωτάω εάν το ιδιωτικό χρέο λαμβάνεται υπόψη στους νέου σχεδιασμού, αυτά τα οποία τον οκτώβριο θα αποφασίσετε κύριε υπουργέ και αν στο πλαίσιο της ε, σχεδιαζόμενης οικονομικής διακυβέρνησης ε, ε, μια νέα ερμηνεία του συμφώνου σταθερότητα, τρόποι εφαρμογή, το ιδιωτικό χρέο έχει κάποια θέση. αν μπορείτε να μου απαντήσετε στην ερώτησή μου θα είμαι πολύ ευτυχής. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ο υπουργό. Όπως έλεγα, η διαδικασία προχωράει. Συνεδριάζει η ομάδα εργασίας, προχτές μάλιστα συνεδρίασε και θα ξανασυνεδριάσει πριν από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Οπότε είναι πρόημο να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για το τι θα γίνει στο μέλλον, για το κριτήριο του χρέους μέσα στο Σύμφωνο Σταθερότητας βάσει των αποτελεσμάτων της Task Force για την Οικονομική Διακυβέρνηση που θα παρουσιάσει την έκθεσή της στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου με έγκριση τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που θα ξεκινήσει ανάλογα με την περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για το ιδιωτικό χρέος. Thank Σας ευχαριστούμε. Έχουμε τώρα ερωτήσεις για το συγκεκριμένο. Δεν έχουμε μάλλον επερωτήσει για το συγκεκριμένο αυτό ερώτημα. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο από την κυρία Τσίκαου. Επανεξέταση του δικτύου Τέντη. Παρακαλώ, Υπουργέ. Μετά από τη δημοσίευση της Επιτροπής ε, μιας πράσινης βίβλου για την επανεξέταση των πολιτικών για καλύτερη ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών ε, δικτύων ε, ε, μεταφορών στα πλαίσια της κοινή πολιτικής μεταφορών, τον Ιούνιο του 2009 υιοθέτησε το ε, Συμβούλιο κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν πρόταση στα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα με στοιχεία σχετικά με τα TEN-T. Υπάρχει η ιδέα του σχεδιασμού σε δύο επίπεδα. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε ένα πρώτο βάθρο κατά κάποιο τρόπο για τις οδικές μεταφορές, για τις εσωτερικές πλωτές ε, επίσης που είναι κάτι που απορρέει από τα διάφορα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και μετά θα έχουμε ένα κεντρικό δίκτυο το οποίο θα δημιουργήσει πραγματικά ευρωπαϊκές προοπτικές και θα έχει να κάνει με την συστημική διασταύρωση των ε, πόρων με ιδιαίτερη προσοχή στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται στις μεταφορές. Υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί δεν ακούγονται αγγλικά στην διερμηνία και από ό,τι φαίνεται ούτε λιθουανικά λέει η πρόεδρος. Έχουμε κάποιο πρόβλημα λοιπόν. Τώρα είναι εντάξει. Συγγνώμη που σας διάκοψα κύριε Υπουργέ. Έλεγα λοιπόν ότι τον Ιούνιο που μας πέρασε το Συμβούλιο σημείωσε τις πληροφορίες που έδωσε η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των ε, ημερίδων της ετήσιας διπουργικής συνάντησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που έλαβε χώρα στη Σαραγώσα. 8 και 9 Ιουνίου. Οι συζητήσεις που έγιναν είχαν σαν αντικείμενο τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε το πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογή των μελλοντικών δικτύων και πώς θα κινητοποιήσουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά πόρους. Έγινε και διαβούλευση με το κοινό από πλευράς της Επιτροπής και έτσι καθορίστηκαν κριτήρια και προϋποθέσεις για το σχεδιασμό σε σφαιρικό και σε κεντρικό επίπεδο. Οι διαδικασίε θα ολοκληρωθούν στι 15 Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα τη διαβούλευση αυτή θα παρουσιαστούν στην Οικονομική Δημοσιονομική Επιτροπή τη 30 Σεπτεμβρίου. Οι επιλογές σχεδιασμού θα συζητηθούν δίμερο, δηλαδή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και πολυμερός στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών αρχές του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει μια μελέτη αξιολόγησης για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών και η πρόταση των κατευθυντήριων γραμμών αναμένεται για τον Ιούνιο του 2011 πριν από την παρουσίαση της πρότασης αυτής και λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση που γίνεται αυτή την εποχή με το κοινό και επειδή θα υπάρξουν και διμερός και πολυμερός διαβουλεύσεις ε, για τα τέλη του 2010, η Βελγική Προεδρία δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο για να προχωρήσει η επανεξέταση του δικτύου TEN-TAF. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ένας από τους ε, στόχους ε, επανεξέτασης ε, της συμφωνίας TNT είναι η υπάρχουσα υποδομή να προσαρμοστεί και σε δίκτυα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις όμορες χώρες. Θα υπάρξει μια ονομαζόμενη ενδιάμεση αναθεώρηση και εμείς θα κληθούμε να καταθέσουμε τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να έχουμε ένα μελλοντικό προγραμματισμό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η συνόρωτησή μου είναι σημαντική. Ο Υπουργός. Η προβληματική στην οποία αναφέρεστε σίγουρα είναι σημαντική και θα αποτελέσει μέρος ε, των συζητήσεων και των προοπτικών που θα αποφασιστούν έτσι ώστε να προσαρμοστούν ανάλογα τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, έχουμε δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις για το ίδιο αυτό θέμα. Μαζί, θα τις ακούσουμε τη μία μετά την άλλη και μετά θα απαντήσετε. Ε, κύριε Σουάντσεφ πρώτα. Ο κύριος Χουντής, Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μόλις πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τα θέματα μεταφορών και τουρισμού, όπου ανέφερε ότι στο πλαίσιο των περικοπών και των δαπανών που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα λόγω του Μνημονίου Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να διακόψει μια σειρά σιδηροδρομικών γραμμών που αποτελούν τμήμα του δικτύου TEN-T και για τι οποίε πρόσφατα δόθηκε χρηματοδοτική ενίσχυση για τον εξυγχρονισμό του από τα διορθωτικά ταμεία. Επειδή αυτή η απόφαση αντιβαίνει για λόγου περιβαλλοντολογικού, για λόγου μείωση των τροχαίων, και παραβίαση του κανονισμού της ευρωπαϊκής ένωσης θα ήθελα να ρωτήσω αν το συμβούλιο προτίθεται να εξετάσει τις καταγγελίες που κάνει ο πρόεδρος της επιτροπής και αν προτίθεται να ζητήσει να ανακληθεί μια τέτοια απόφαση. Κύριε Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ερώτημα που ετέθη η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη αυτών των δικτύων είναι πάρα πολύ σημαντική, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όμως η εξέλιξη πρέπει να είναι συνεπής και αυτό επίσης είναι πολύ δαπανηρό. Η δική μου λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής. Στον προπολογισμό του 2014-2020 Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα να αυξηθούν τα κονδύλια για αυτά τα δίκτυα, να αυξηθούν περαιτέρω. Ο κύριος Υπουργό. Στην πρώτη ερώτηση για την μείωση των δυνατοτήτων της Ελλάδας να επενδύσει στα δίκτυα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για το θέμα αυτό μπορούμε να μάθουμε. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω συγκεκριμένα για το με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιδράσουμε στη μείωση της δυνατότητας που έχει η Ελλάδα. Θα έρθω σε επαφή με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντως για να δω πώς μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Τώρα, για την ανησυχία για τη συνοχή και για τα οικονομικά μέσα που πρέπει να διατεθούν, εδώ ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κοιτάξει λίγο την έννοια των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020. Εσείς θα αποφανθείτε επίσης για το θέμα αυτό, ανάλογα βάσει μάλλον της αρχής για τη συναπόφαση στα δημοσιονομικά. Βασίζομαι λοιπόν σε εσά για να βάλετε στην ατζέντα των μελλοντικών συζητήσεων για τον προπολογισμό, ώστε να ληφθεί υπόψη η συνοχή αυτή με τους στόχους των μεταφορών. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, Πρόεδρος. Τώρα περνάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι του κυρίου Παπα-Νικολάου και έχει να κάνει με την αξιολόγηση της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ όταν μπορείτε. Στα συμπεράσματά του τη 30 Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο επενθύμησε ότι η ανοιχτή μεθόδο συντονισμού συνεισέφερε στην καλή λειτουργία της αγοράς εργασίας αλλά και ε, της κοινωνικής ε, συμπερίληψης των ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο. Και στο μέλλον η μέθοδος αυτή θα είναι χρήσιμη. Βέβαια, χρειάζεται αποτελεσματικός έλεγχος των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση που θα υιοθετηθούν προσεχώς από το Συμβούλιο μετά την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στο κάτω-κάτω σήμερα αποφασίσατε γι' αυτήν και που είναι πολύ σημαντική για το Συμβούλιο στα πλαίσια της νέας διακυβέρνησης, κάτι το οποίο θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πέρυσι, εξάλλου, όταν το Συμβούλιο υιοθέτησε ένα νέο πλαίσιο στατικής σημασίας για ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι νέες χώρες μέλη ε, παραδέχτηκαν ότι οι στόχοι έχουν ως προϋπόθεση τη λειτουργία της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Συνεχίζουν λοιπόν να στηρίζουν τη μέθοδο αυτή, η οποία είναι όντως ιδιαίτερα χρήσιμη στους τομείς που έχουν να κάνουν με τις εθνικές αρμοδιότητες. Η πρόσφατη μεικτή έκθεση για το 2010 του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας Εκπαίδευση κατάρτιση 2010 επιστήνει την προσοχή στις σημαντικές πρόοδους που διαπιστώθηκαν χάρη στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Προς την ίδια κατεύθυνση, στα συμπεράσματα του, του Ιουνίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέστησε την προσοχή μας στο πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι συζητήσεις που γίνονται για τη στρατηγική 2020 και ότι εκεί πρέπει να ληφθεί υπόψη η μέθοδος αυτή, η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού και στον τομέα της προστασίας και μείωσης ε, της απομόνωσης. Οι δυνατότητες είναι μεγάλες στα πλαίσια της Αττικής 2020 για την εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού. Θέλουμε μείωση της φτώχειας, ενίσχυση των κοινωνικών διαστάσεων και στην κατευθυντήρια γραμμή 10, στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών ε, Κοινωνικών Υποθέσεων 9 Ιουλίου, η Πρόεδρος ζήτησε από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερο την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Μάλιστα στο ψήφισμα του Νοεμβρίου το 2009 που μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία όσον αφορά την ε, νεολαία σε ένα πρόγραμμα 2010-2018, το Συμβούλιο έχει ήδη θέσει τις βασικές αρχές που πρέπει να ισχύουν σε όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με την νεολαία. Και αυτό μέσα στα πλαίσια μια ανανεωμένης ανοιχτή μεθόδου συντονισμού. Έτσι, η Προεδρία θα οργανώσει 14 Σεπτεμβρίου μία διάσκεψη και το Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα ξανασυζητήσει το θέμα αυτό και θα καταλήξει σε συμπεράσματα για την απασχόληση και για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. κύριο Κύριος Παπα-Νικολάου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Θα ήθελα όμως να μου διευκρινίσετε τα εξής. Πράγματι, η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού σε κρίσιμου τομεί του αναφέρατε κι εσεί η εκπαίδευση η απασχόληση η κατάρτιση τα θέματα νεολαία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μα στα πλαίσια μάλιστα και τη επικουρικότητα ε, και των αρμοδιοτήτων που έχει η ευρωπαϊκή ένωση. ερωτώ θα μπορούσαμε να έχουμε κατά καιρού κάποια πορίσματα αυτή τη μεθόδου για την ανταλλαγή των απόψεων προκειμένου και εμεί σε πολιτικό επίπεδο να έχουμε ενημέρωση. και δεύτερον το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πώ θα μπορούσε πιο ενεργά να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου και εμεί να τα αναδείξουμε περισσότερο. σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Στο τελευταίο τμήμα της απάντησής μου, το λέω λίγο πολύ, αλλά βέβαια τα συμπεράσματα της 21ης Οκτωβρίου του Συμβουλίου δηλαδή τότε θα σας δοθούν πολύ συγκεκριμένα. Θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για τα θέματα της απασχόλησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα ενημερωθείτε, γι' αυτό θα είναι στη διάθεσή σας. Νομίζω ότι υπάρχει άλλη μια συμπληρωματική ερώτηση από την κυρία Μπλικιπιτσούκα. Κοιτάξτε, σε σχέση με τη μέθοδο της, ε, την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και τη σημασία της, φέτος έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος καταπολέμησης της φτώχειας και είναι σύμπτωση το ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε έντονο κοινωνικό αποκλεισμό. Πρέπει λοιπόν ε, να καταπολεμήσουμε την φτώχεια. Εσείς λέτε ότι θα υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ότι θα μάθουμε από τις σκανδιναβικές χώρες, γιατί οι χώρες αυτές ε, μαθαίνουν από την καταπολέμηση της φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θεωρείτε λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η φτώχεια στις χώρες της Βαλτικής συντονισμός και αμοιβαία ε, εκμάθηση καλών πρακτικών είναι θετικά στοιχεία. Εσείς υπογραμμίσατε μια από τις πτυχές προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι για τα κοινωνικά ζητήματα και ιδίως για την ανάπτυξη. Η απασχόληση, η καταπολέμηση τη φτώχειας προφανώς είναι τα καταξοχήν θέματα για το 2010 και κυρίως η πολιτική της ε, ενεργού συμμετοχή. Δεν θέλουμε μόνο να μειώσουμε την ε, φτώχεια, αλλά να αυξήσουμε και την προσφορά εργατικού δυναμικού, να μεταρρυθμίσουμε ενδεχομένω τα συνταξιδοτικά συστήματα. Όλα αυτά μπορεί να αυξήσουν και το ποσοστό απασχόληση και να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των ε, δημόσιων νομικών ε, και ιδίω για τον τομέα τη υγειονομική περίθαλψη. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι το 2010, έτο αφιερωμένο στην καταπολέμηση τη φτώχεια, θα μπορέσουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε τον συντονισμό και την αμοιβαία αυτή εκμάθηση και ανταλλαγή εμπειριών. Ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο ερώτημα από τον κύριο Χουντή. Μνημόνιο αμοιβαία Κατανόησης ε, Ελλάδα, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Και ταυτόχρονα το φαινόμενο τη έκρηξη του πληθωρισμού. Το Συμβούλιο τόνισε επανειλημμένο στα διαφορετικά μακροχρόνια προβλήματα της άμεσης οικονομίας και αυτό στις διάφορες διαδικασίες πολυμερούς ε, οικονομικής ε, επαγρύπνησης. Για τα υπέρμετρα χρέη, το 2010 το Συμβούλιο πρότεινε στην Ελλάδα να, να λάβει ένα σύνολο μέτρων προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργία των αγορών προϊόντων και το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις προκειμένου να τονώσει την ε, ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την απασχόληση. Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και το ρυθμό απορρόφησης των ιδιωτικών ταμείων της και κορνελίων της Ένωσης και να διορθώσει το ε, μεγάλο έλλειμμα στον προπολογισμό τη, καθώ και να εξηγειάνει μακροπρόθεσμα τα δημοσιονομικά τη. Η Ελλάδα λοιπόν υπέβαλε την πρώτη έκθεση για την υλοποίηση των ε, μέτρων αυτών στι 16 Μαρτίου και έπειτα τη δεύτερη τον Μάιο. Τον Ιούνιο η Επιτροπή και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο πραγματοποίησαν μια προκατακτική ανάλυση των συμπερασμάτων στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξη για τη σταθερότητα με μια αξία 110 δι ευρώ που συνέβαλαν από κοινού τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνέ Ταμείο προς την Ελλάδα. Η ανάλυση αυτή ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο, Όμω το Συμβούλιο δεν έλαβε επισήμω την τελική έκθεση της Επιτροπής, διότι η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για τα πορίσματα, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της συγκεκριμένη ανάλυση. Βάσει της αξιολόγηση της Επιτροπής, η εξέλιξη της οικονομίας είναι σύμφωνη με τους στόχους που έχει θέσει το πρόγραμμα αυτό, συνοδεύοντας τους στόχους τους μηχανισμούς σταθερότητας, ε, ενώ η αύξηση του πληθωρισμού δείχνει ότι δεν υπάρχει ατελής λειτουργία της αγοράς προϊόντων. Το Συμβούλιο εξετάζει προσεκτικά την κατάσταση και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα εφόσον χρειαστούν, προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές να ε, βελτιώσουν την ε, οικονομική ανάπτυξη και να ε, ακολουθήσουν μια υγιή δημοσιονομική πολιτική. Βάσει της αξιολόγηση της Επιτροπής, η εξέλιξη της οικονομίας συμπίπτει με τις προβλέψεις του προγράμματος ε, και του στόχου σταθεροποίηση, όμως η αύξηση του ποσοστού του πληθωρισμού δείχνει ότι είναι ατελή η λειτουργία των αγορών όπως σας προείπα. Και η δημοσιονομική κατάσταση είναι ένα στοιχείο που θα παρακολουθεί προσεκτικότατα συνεχώ το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, φοβάμαι ότι δεν απαντήσατε στο ερώτημα που σας έθεσα τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στην ελλάδα λόγω του μνημονίου τη διαδικασία την οποία μου περιγράψατε μνημονίου Διεθνού νομισματικού ταμείου και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχιζοφρενικά. από τη μια πλευρά προκειμένου να εισπραχτούν κρατικά έσοδα επιβάλλονται φόροι φόροι που δεν μπορούν να εισπραχτούν διότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλο εισόδημα οι μικρέ επιχειρήσεις το ίδιο και ενώ μιλούν για αποπληθωρισμό σχεδιάζουν νέα φοροεισπρακτικά μέτρα με αύξηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αύξηση της φορολογίας του πετρελαίου θέρμανσης. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι, από τις πληροφορίες που έχω, στο χτεσινό ΕΚΟΦΗΝ ενθαρρύνθηκε η Ελλάδα να πάρει νέα φοροεισπρακτικά μέτρα που σημαίνει έκρηξη του πληθωρισμού. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, το ΕΚΟΦΗΝ έχει συζητήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει πέρα από τα φοροεισπρακτικά μέτρα, διορθωτικά μέτρα για να μην έχουμε έκρηξη πληθωρισμού στην Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση για το τι αποφάσισε το ΕΚΟΦΗΝ πριν από λίγο. Αλλά ε, πολλές φορές μέχρι τώρα έχει ασχοληθεί το Συμβούλιο με το πρόβλημα της Ελλάδας και με την ε, πολυμερή εποπτεία και βάσει τα στρατηγικής απασχόλησης της Λισαβόνας για την απασχόληση, τις συστάσεις του το Συμβούλιο για την ενημέρωση των κατευθυντηρίων γραμμών των κρατών μελών είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερες προσπάθειες για να μην υπάρχουν ε, μακροπρόθεσμες ανισορροπίες και διαρροτικά προβλήματα στην οικονομία της. Και το Συμβούλιο συστήνει στην Ελλάδα να αυξήσει τον ανταγωνισμό στον τομέα των ε, επαγγελματικών υπηρεσιών και τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, να χρησιμοποιήσει διαφορετικά ε, τα, τα ταμεία πιο αποτελεσματικά και να φροντίσει η ελληνική διοίκηση να πάρει μέτρα υπέρ τη αγορά τη απασχόληση στα πλαίσια μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ευελιξία και την ασφάλεια. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι ελληνικέ αρχέ επιβεβαίωσαν ότι έδωσαν την προτεραιότητα σε πολλέ διεθνωτικές μεταρρυθμίσει που σχεδίασαν σε διάφορου τομεί και κλάδου. Ε, Ξέροντα τι δυσκολίε που δημιουργούνται βέβαια στη χώρα εξαιτία αυτών των μέτρων. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Έχω και άλλη συμπληρωματική επί του θέματος από τον κύριο Παπα-Νικολάου. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Χουντής, ο πολύ καλός συνάδελφος, στην ερώτησή του αναφέρει ότι ο πληθωρισμός τον Ιούλιο ήταν 5,4. Τον Αύγουστο ανακοινώθηκε ότι είναι 5,5. Και φαίνεται ότι με τη λήψη νέων μέτρων σε είδη λαϊκής κατανάλωσης όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο συνάδελφος προηγουμένως ο πληθωρισμός είναι πάρα πολύ δύσκολο να μειωθεί και την ίδια στιγμή ξανά συζητάμε για μέτρα όπως μας λέτε στα πλαίσια του συμβουλίου πάλι για νέους φόρους και ρωτώ, μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα πιο συγκεκριμένα έχουμε τόσο από την πλευρά του Συμβουλίου, της Ευρώπης, του Μηχανισμού Στήριξης, όσο όμω και από την πλευρά τη Ελλάδας. Έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ο πληθωρισμός ε, δεν είναι αυξανόμενος και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και πρέπει να υπάρξει ισορροπία αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ως μέλος της Ευρωζώνης η Ελλάδα έχει την ίδια ευθύνη που έχουν και άλλες χώρες μέλη για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Η οικονομική πολιτική λοιπόν της Ελλάδας εντάσσεται στα ίδια πλαίσια όπως και εκείνη των άλλων χωρών και δημιουργεί τις ίδιες ανησυχίες όπως γνωρίζουμε και από το Σύμφωνο σταθερότητα. Η χώρα λοιπόν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο για να μειωθεί ο κίνδυνος να μην μπορεί να λειτουργήσει καλά η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Thank you, Minister. We now move on... Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Συνεχίζουμε και περνάμε στην επόμενη ερώτηση τώρα που είναι της κυρίας Άντρη και έχει να κάνει με τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας όσον αφορά τον ΟΗΕ και τα όργανα του. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Στα πλαίσια της 65ης ε, συνέλευσης του ΟΗΕ, το Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2010 ενέκρινε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να επενθυμίσω ότι η άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας είναι ο ύπατος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας να ασχοληθεί με το θέμα αυτό την εκπροσώπηση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ μεταξύ άλλων. Οι προτεραιότητες είναι να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί και το Συμβούλιο δουλεύει υπέρ ενό ενισχυμένου πολυμερού συστήματος. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διαφάνεια, την υπευθυνότητα, την αποτελεσματικότητα των ΗΕ. Δεύτερη προτεραιότητα θα είναι να συνεισφέρουμε στην ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει την προβολή των θέσεών της και να συνεισφέρει στη διαχείριση κρίσεων μέσα από τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων το Συμβούλιο Ασφαλείας για παράδειγμα. Τρίτη προτεραιότητα θα είναι το περιβάλλον και η αηφόρος ανάπτυξη. Και αυτό προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Τέταρτη προτεραιότητα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα από εκείνου που πιο αποφασιστικά ε, στήριζαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και που συμμετέχουν στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενθαρρύνει δραστήρια τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να συμπεριληφθούν σε όλες τις δράσεις του ΟΗΕ και να φροντίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνδέονται άρρηκτα με τους άλλους στόχους του ΟΗΕ, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Τέλος, πέμπτη προτεραιότητα είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ και αυτό προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα αλλά και η αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος. Όσον αφορά την μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Human Rights Council Review, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στις ε, ε, επίσημες και τις άτυπες διαβουλεύσεις και θέλουμε η Τρίτη Επιτροπή να ενισχύσει τις αρμοδιότητες της που έχει αρμοδιότητες σε θέματα προδιαγραφών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να διατηρηθούν οι αρμοδιότητες αυτές. Όσον αφορά τώρα το θέμα τη διπλωματική εκπροσωπηση από 1 Δεκεμβρίου 2009 όλε οι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής στο εξωτερικό είναι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και στη Γενέβη η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Γραφείο Σύνδεση τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που υιοθέτησε ε, τρόπους λειτουργίας προσωρινά μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Thank you. Παρακαλούμε, κύριε Αντρέκενε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την απάντησή σας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση για το πώς ακριβώς ε, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη και αυτό υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, μετά από πολλές συζητήσεις για τις προτεραιότητες <coughs> και σε σχέση με την αναθεώρηση του Συμβουλίου Περιανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Βελική Προεδρία και είπα της εκπρόσωπος πρέπει να διασφαλίσουν ότι τώρα πλέον θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία ε, για να εξεταστεί η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα κράτη-μέλη. Επίσης πρέπει να υπάρχει αρχηγικό πνεύμα, κυρίως στο ψήφισμα για την, ε, για την θανατική πυκνή και για, την, ε, για το εμπόριο των όπλων. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις δικές σας απόψεις του θέματος. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε. Έχετε κάποια σχόλια για αυτά τα θέματα. Ίσως να περάσουμε... Ε, α, εντάξει, ωραία. Μισό λεπτό. Απλώς να σας πω ότι το Βέλγιο προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και είναι και μέλος του Συμβουλίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Βεβαίως θα φροντίσει να επαγρυπνεί και να λάβει υπόψη τις μέρημνες που αναφέρατε. Ευχαριστούμε. Έχω μια επερώτηση από τον κύριο Ρούμπικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα είχαμε μια αρκετά έντονη συζήτηση όπου ε, ζήτησαμε εξηγήσει ε, από το Συμβουλίο για τις Εξοικονομήσεις ε, στο 2011. Θα το στηρίξουμε το Συμβούλιο και κατά τα άλλα η διπλωματική υπηρεσία που είναι υποσύσταση συζητήθηκε ενδελεχώς. Πιστεύετε εσείς ότι στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να αναλυθούν προσπάθειες έτσι ώστε οι θέσεις ε, να καλύπτονται αποτελεσματικότερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ομιλεί με μία φωνή. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια τα οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σε άλλους τομείς. Η Βελγική Προεδρία είναι πρόθυμη να ε, καταθέσει προτάσεις ε, εξοικονόμησης που θα υπηρετούν αυτό το στόχο ε, της αποτελεσματικότερης εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός. Εφ' εξής, προβλέπονται διάφορα μέτρα ενίσχυσης και στην Νέα Υόρκη και στην Γενέβη, αλλά μέσω του ερωτήματό σα να σα επιστήσω το γεγονό ότι θα πρέπει να θέσουμε σε άμεση λειτουργία και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Εδώ έχει και το Κοινοβούλιο ένα ρόλο να διαδραματίσει, ιδίω ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά και την άμεση ίδρυση και λειτουργία αυτή τη υπηρεσία. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση από τον κύριο Aylward αφορά την ενίσχυση της επικοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Πιθανές επιλογές» για το διάστημα μετά το 2010 και σε ό,τι αφορά του προσανατολισμού και του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βιοπικιλότητα, το Συμβούλιο ενέκρινε στι 15 Μαρτίου 2010 συμπεράσματα με τον τίτλο Βιοπικιλότητα μετά το 2010, όραμα και στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνέ επίπεδο. Επίση, διεθνέ καθεστώ πρόσβαση και ε, κατανομή των πλέον εκτιμάτων, των ωφελών. Σε αυτή τη δήλωση το Συμβούλιο επισημαίνει την ανησυχία του σε σχέση με το ότι στόχοι για το 2010 και ω προ την βιοπικιλότητα δεν επετέφθησαν ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο παγκόσμιο. Η απώλεια της βιοπικιλότητας εξακολουθεί με ρυθμό απαράδεκτο και επιφέρει συνέπειες οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές πολύ δεσμενείς. Εδώ λοιπόν πρέπει να, να υπογραμμιστεί ότι οι στόχοι αυτοί παίζουν καθοριστικό ρόλο, διότι ε, αρχικά είχαν επιτρέψει την λήψη σημαντικών μέτρων για την προστασία τη βιοποικιλότητας. Επίση, συνοδεύονται από ένα μακροπρόθεσμο όραμα, βάσει του οποίου το 2050 η επικοινότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπηρεσίες για τα οικοσυστήματα που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το συνολικό ζωικό κεφάλαιο, θα προστατεύονται, θα προωθούνται και θα αναβαθμίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της βιοπικιλότητα και της συμβολής της, της καθοριστικής συμβολής την ε, ευημερία του ανθρώπου, καθώς και την οικονομική ευημερία οι καταστροφικές συνέπειες από την απώλεια επικοινότητας θα αποφεύγονταν και αυτό είναι ένα από του πρωταρχικού στόχου προκειμένου να, να ανακόψουμε την απώλεια επικοινότητα και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2020. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε δυνατό τρόπο προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην μείωση της ε, ε, απώλειας σε επίπεδο πλανήτη. Ω προ τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία και την ενίσχυση τη βιοπικιλότητα, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η καταστροφή, ο κατακαιρματισμός και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων είναι από τα στοιχεία που περισσότερο πλήττουν τη βιοπικιλότητα. Προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση λοιπόν των οικοτόπων, το Συμβούλιο έχει προβλέψει πρόγραμμα για την προστασία των εδαφών, την καταπολέμηση της υπερεκμετάλλευσης, την προστασία των φυσικών πόρων, τα επιθετικά εξωτικά είδη, τα είδη που απελούνται με εξαφάνιση και την ρήπανση. Επίσης, οι κλιματικές αλλαγές μπορεί να επιβαρύνουν κάποιες από τις συνθήκες, όπως τον αριθμό των ε, υποεξαφάνιση ζωικών ειδών. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική Ευρώπη 2020, η αδρή προσανατολισμοί τη Επιτροπή και του Συμβουλίου οδηγούν στο να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη να προβλέψουν μέτρα ώστε οι προκλήσει περιβαλλοντικέ να μετατραπούν σε ωφέλη και να αξιοποιούν κατάλληλα τους φυσικούς πόρους. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στο να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα, το ρόλο της βιοπικιλότητας, τον τόνισε επίσης το Συμβούλιο στα συμπεράσματα του το Μάρτιο του 2010, όταν δήλωσε ότι είναι κατεπήγον να αντιστραφεί η σημερινή τάση για απώλεια της βεπικιλότητας και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και βεβαίως το Συμβούλιο προσυπογράφει στη μακροπρόθεσμο το ευρύτερο αυτό όραμα για τον ορίζοντα του 2050 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τους στόχους του 2020, όπως ορίζονται στα συμπεράσματα που σας προανέφερα από το Συμβούλιο της 15ης Μαρτίου 2010. Thank you very much, Minister. Ευχαριστούμε πολύ, είναι απογοητευτικό να ακούμε από τον Υπουργό ότι δεν υπάρχει πρόοδος προκειμένου να πετύχουμε την προστασία της βιοποικιλότητας. Τώρα με τα μέτρα που θέλουμε να πάρουμε μπορούμε να βελτιώσουμε την βιοποικιλότητα. Στο μεταξύ το Συμβούλιο τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να ενισχύσει τους γεωργούς, οι οποίοι πρωτίστως έχουν το ρόλο προστασίας της βιοπικιλότητας. Κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι το καλύτερο μέτρο για να προστατεύσουμε την ε, καλή δουλειά στη Γεωργία είναι ακριβώς να τη στηρίξουμε. Και εδώ θέλω να πω στους παρόντες, αν και δεν είναι και πάρει πολύ, πάρα πολύ, στην επόμενη συζήτηση που θα γίνει για αυτό το θέμα, να στηρίξουν με τις δημοσιονομικές αποφάσεις που θα πάρουν την κοινή γεωργική πολιτική. Βασίζομαι σε εσά λοιπόν. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλη συμπληρωματική ερώτηση για αυτό το θέμα. Και έτσι περνάμε στην επόμενη ερώτηση της κυρίας Μαγκίνες που έχει να κάνει με το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας του Σεπτεμβρίου 2010 φέτος. Κύριε Υπουργέ. Ε, κύριε Άουαρτ, έχετε κάτι διαδικαστικό, τι συμβαίνει. Όχι, ο Υπουργός. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, επιτυχίες που πέτυχε όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική για μετά το 2013. 6.000 παρεμβάσεις από το κοινό, διάφορες ομάδες, προβληματισμού, έρευνας κλπ. Το συνέδριο λοιπόν πέτυχε πολύ. Επίσης, οι παρεμβάσεις έδειξαν ότι ολόκληρη η κοινωνία μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι υπόθεση μόνο των γεωργών. Όπως ξέρετε, η διαβούλευση οδήγησε στην διάσκεψη για την ΚΑΠ μετά το 2013 που έλαβε χώρα τον Ιούλιο που μας πέρασε. Οι παρεμβάσεις, οι συζητήσεις τροκιλής ε, τραπέζης και που έλαβαν χώρα αποτελούν πολύτιμο υλικό για να προχωρήσουμε στις αποφάσεις μας. Από την πλευρά του το Συμβούλιο, ξέρετε ότι ε, ο Υπουργός Γεωργίας τα δύο τελευταία χρόνια ε, φρόντισε να γίνει μια δουλειά προβληματισμού με συνεργασία της Γαλλικής, της Τσεχικής, της Σουηδικής και της Ισπανικής Προεδρίας. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία και προσπαθούμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Είναι βασικό η πραγματικότητα της σημερινής ΚΑΠ και οι προκλήσεις της αυριανής ΚΑΠ να εκτιμηθούν σωστά στη συζήτηση που θα γίνει στα πλαίσια ε, του προπολογισμού και των δημοσιονομικών ε, προοπτικών της Ένωσης 2014-2020. Το μέλλον της ΚΑΠ ξέρετε ότι θα αποτελέσει κεντρικό σημείο στις συζητήσεις του άτυπου συμβουλίου που θα λάβει η χώρα 19 με 21 Σεπτεμβρίου στο Βέλγιο. Ο κύριος Δεκάστρο, πρόεδρος της Επιτροπής σας Γεωργίας, ε, προσεκλήθη να συμμετάσχει στην συνάντηση αυτή και να συμμετάσχει στις άτυπες συζητήσεις. Η Προεδρία φάντως φέτος το καλοκαίρι ε, συζήτησε τα αποτελέσματα της συνάντησης του Ιουλίου και θα καταλήξει μέσα στις δύο επόμενες ημέρες. Ο απολογισμός πάντως της Προεδρίας και στον οποίο θα εμβαθύνουμε περισσότερο τις επόμενες μέρες, επιβεβαιώνει ότι οι στόχοι της ΚΑΠ είναι σωστοί, έτσι όπως αυτοί αναφέρονται και στην συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή να έχουμε ασφαλή και ποιότητα στρόφιμα για τον Ευρωπαίο πολίτη, να έχουμε μια βιώσιμη γεωργία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και ε, το, τις τοποθεσίες, το τοπίο και ότι άλλο έχει σχέση με τα προηγούμενα. Πάντως ο απολογισμός της Προεδρίας επιβεβαιώνει επίσης την πρόσθετη αξία της κοινή γεωργική πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη σημασία που έχει η ΚΑΠ στα πλαίσια της Στρατηγική Ευρώπη 2020. Οι επόμενες συζητήσεις θα οδηγήσουν τον Οκτώβριο σε μια τελευταία συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ στο Συμβούλιο Γεωργίας. Έτσι το Συμβούλιο θα έχει συνεισφέρει όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεγάλο βαθμό στη διαδικασία προβληματισμού. Είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης συζητάει το έργο του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σίγουρα θα κάνει ό,τι προσπάθειες χρειάζονται για να παρουσιάσει ανακοίνωση η οποία θα υποστηριχθεί από τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Όταν θα είναι στη διάθεσή μας η ανακοίνωση αυτή, θα ξεκινήσει η συζήτηση στο Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις χώρες Μερκοσούρ, εδώ θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι φυσικά και ξέρω πόσο μεγάλη οικονομική σημασία έχει η συμφωνία αυτή, αλλά η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι Υπουργοί Γεωργίας ε, πρέπει να ξέρετε ότι επίσης συμφωνούν. Αλλά ξέρουν ότι είναι μια συμφωνία η οποία λοχεύει κινδύνους για κάποιους ευαίσθητους κλάδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μάιο που μας πέρασε το Συμβούλιο σημείωσε τις ανησυχίες που εξέφρασαν διάφορα κράτη-μέλη σε ένα κοινό σημείωμα. Υπενθυμίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τηρεί την εντολή που έχει για διαπραγματεύσεις. Εξάλλου το Μάιο ο Επίτροπος Ιόλος είπε στο Συμβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φροντίσει οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες Μερκοσούρ να είναι συμβατές με την κοινή γεωργική πολιτική και με τα βασικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Εν κατακλείδη, θέλω να υπογραμμίσω ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συζητήσεις που γίνονται με τις χώρες Μερκοσούρ μέσω της Επιτροπής για την Εμπορική Πολιτική. Οι επόμενες συζητήσεις θα γίνουν τον Οκτώβριο και σας διαβεβαιώ ότι το Συμβούλιο θα φροντίσει να τηρηθεί πλήρως η εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Η απάντηση ήταν ε, λεπτομερής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, κυρίως αυτά που είπατε για το Μερκοσούρ και πράγματι ελπίζω οι ε, Κομισιόν και το, Συμβούλιο να καταγράψουν τις δικές μας τις ανησυχίες. Στην απάντησή σας στον συνάδελφό μου για την βιοπικιλότητα και τα σχόλιά σας για τον γεωργικό ε, προπολογισμό με οδηγούν στο να ε, ζητήσω και την άποψη του ε, Συμβουλίου. Προτίθενται του χρόνου να περικόψουν τον προπολογισμό και αυτό δεν είναι καλό ιονό για τον επόμενο προπολογισμό για τη Γεωργία. Ο κύριος Υπουργό έχει το λόγο. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να μειώσουν το σύνολο του προπολογισμού για τον χρόνο. Εξ όσων γνωρίζω όμως εγώ, η συμφωνία στο Συμβούλιο δεν ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Κατά βάση πιθανότητα θα ακούσατε χθε τον Βέλγο Υπουργό, που είναι υπεύθυνο για τον προπολογισμό, να παρουσιάζει τα του προπολογισμού για το 2011 και θα ακούσατε ποιε είναι οι προοπτικέ οι δημοσιονομικές για το 2011. Μόλις ξεκίνησαν οι συζητήσεις με το Κοινοβούλιο. Εγώ δεν με τη δική σας την παρουσίαση για το πώς εξελίσσεται ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Ο κύριο Ρούμπικ. Κυρία Πρόεδρε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι κατά πόσον ο προπολογισμό 2011 συζητείται αυτή τη στιγμή και το Συμβούλιο πρότεινε από κοινού με την Κομισιόν τα κονδύλια για το πρόγραμμα ανταγωνισμού και καινοτομιών, ε, το πρόγραμμα το ICT ε, και ένα άλλο πρόγραμμα την επιχειρηματικότητα αλλά και το έβδομο ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο όλα αυτά να συγχωνευθούν. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια ακριβώς ε, είναι η άποψη Προεδρίας επ' αυτού. Ο κύριος Αλγούτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας κατά νου την απόφαση της ε, Κομισιόν να ξεκινήσει και πάλι τις συζητήσεις για το Μερκοσούρ, μήπως μπορείτε να μας πείτε κατά πόσον το Συμβούλιο σκέπτεται τις ε, καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτή η απόφαση για τους ε, Ευρωπαίους ε, γεωργούς, κυρίως της δικής μου της χώρας, που κατά 90% εξαρτώνται από τις εξαγωγές βοηδών, εξαγωγές που γίνονται με βάση αυστηρότατα κριτήρια, κριτήρια που δεν ισχύουν στις χώρες Μερκοσούρ. Ο κύριος Υπουργό έχει το λόγο. Για την πρώτη ερώτηση σας παραπέμπω στη γενική παρουσίαση που προς στιγμήν έγινε για τον προπολογισμό. Ε, υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία γνωρίζω ότι είναι προσφύλη για το Κοινοβούλιο όπως για την ε, καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία αλλά μόλις ξεκινάει ο αγώνας έχετε από την 1η Δεκεμβρίου κάθε ευκαιρία την περασ... του περασμένου έτου μάλιστα, κάθε ευκαιρία για να τροποποιήσετε τον προπολογισμό τη επόμενη χρονιά. Σα παραπέμπω λοιπόν στη δημοσιονομική συζήτηση για να δείτε ποια είναι η έμφαση που θέλουν να δώσουν σε κάποιε προτεραιότητε οι ευρωβουλευτέ σε σημεία του προπολογισμού. Τώρα για τη Μερκοσούρ, όπω σα είπα, η Προεδρία είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη και συμμερίζεται τι ανησυχίε τη Επιτροπή Γεωργία και ανάπτυξη τη υπαίθρου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σα είπα ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών η Επιτροπή παρέμεινε πιστή στην διαπραγματευτική τη εντολή και ότι όλα τα θετικά ε, στοιχεία ε, που θα συζητηθούν στι διαπραγματεύσει αυτέ, που θα ωφελήσουν τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η προώθηση, η μεγαλύτερη πραγματοποίηση των ε, γεωργικών προϊόντων από την Ευρώπη και τι γεωγραφικέ ενδείξει, όλα αυτά είναι στοιχεία που θα τα προωθήσουμε. Thank you, Minister. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα στο, στην επόμενη ερώτηση που αφορά τις προοπτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Βαλκανικών κρατών. Ο στόχος της πολιτικής μας απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια είναι η σταθερότητα στην περιοχή. Εξάλλου θέλουμε να υπάρξει στις χώρες της περιοχής ειρήνη και ευημερία, όπως επίσης και σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που είναι ένα πλαίσιο που οδηγεί στην δυνατότητα προσχώρησης των χωρών αυτών και αυτό ώστε σταδιακά να δούμε τις προοπτικές προσχώρησης των χωρών αυτών. Είναι σημαντικό στοιχείο η προοπτική αυτή γιατί τη και το μέλλον της περιοχής. Ε, προχωράει σύμφωνα με την Θεσσαλονίκη, την ατζέντα της Θεσσαλονίκης και λαμβάνονται υπόψη προϋποθέσεις οι οποίες είναι ισότιμες αλλά και αυστηρές. Το Συμβούλιο λοιπόν έχει επαναλάβει ξανά και ξανά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Βαλκανίων και το είπε και στα πλαίσια του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου μετά από τη συνεδρίαση στο Σαράγεβο 2 Ιουνίου που μας πέρασε. Με τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει έξι συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με χώρες από την περιοχή. Τέσσερις έχουν αρχίσει ήδη να ισχύουν. Από τον Οκτώβριο ε, πρότεινε η Επιτροπή να ξεκινήσουν ε, διαπραγματεύσεις με την ε, και με την Κροατία ξέρετε ότι έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις και βρίσκονται τώρα στο τελικό στάδιο. Πολιτικά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι μέσα διαθέτει με την ΚΕΠΑ, με την Βοσνία Ζεγοβίνη και το Κωσυφοπέδιο και με δύο ειδικέ αποστολές στα Σκόπια, στην Πριστίνα και στο Σαράγεβο προχωράει. Η ενίσχυση θα είναι πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ για το 2010 και θα είναι ένα δις το 2013. Η οικονομική αρρωγή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της περιοχής ξεπερνούν τα 13 δις από το 1991 και εφεξής. Όσον αφορά την ημερομηνία προσχώρησης, εξαρτάται από την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεχάγης και των προποθέσεων που έχουν μπει με τις συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης. Ε, συμφωνία σταθεροποίηση και σύμβαση, μετά γνωμοδότηση, μετά υποψήφια χώρα, ε, μετά διαπραγματεύσει για προσχώρηση και μετά προσχώρηση. Το Συμβούλιο λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, περιμένει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Αλλά είναι στα χέρια των κυβερνήσεων της περιοχής να συνεχίσουν και να εντατικοποιήσουν το ρυθμό με τον οποίο γίνονται οι μεταρρυθμίσεις, κάτι το οποίο είναι βέβαια μια μεγάλη πρόκληση για την περιοχή οι χώρε πρέπει να κάνουν περισσότερε προσπάθειε για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει επίση να ενισχυθεί ο διοικητικό του ιστό και να φροντίσουν να διακανονιστούν τα σε κρεμότητα θέματα. Στόχο τη διαδικασία σταθεροποίηση και σύνδεση δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο εφόσον οι κυβερνήσει και λέει τη περιοχή δραστηριοποιηθούν με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα. Το μέλλον τη περιοχή εξαρτάται τελικά από ε, τους λαούς και τις κυβερνήσεις, από την ε, πολιτική καλής γυτνίασης, από το διακανονισμό των ε, διμερών διαφορών που υπάρχουν στην περιοχή. Οι πολιτικές αυτές είναι πολιτικές που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή και στις οποίες επιμένουμε από το 1995. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο 14 Ιουνίου που μας πέρασε ζήτησε από τις διαφερόμενες χώρες να λύσουν ό,τι διαφορές έχουν με τις γειτονές χώρες. Θέλω να ολοκληρώσω υπενθυμίζοντας ότι το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2009 ε, συμφώνησε για ελευθέρωση του συστήματος θεωρήσεων για τρεις χώρες της περιοχής, όπως επίσης για την Αλβανία και τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ελπίζω να πάρουν την ε, τελική απόφαση ακόμα φέτος. Τέλος, όσον αφορά ε, τις επιπτώσεις της διεύρυνσης τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα για τι δημοσιονομικέ προοπτικές 2014-2020, το Συμβούλιο δεν μπορεί τώρα να εκφραστεί γιατί περιμένει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστούμε πολύ. κύριε Τζανάκη. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που η συζήτηση ε, διεξάγεται τόσο ήπια, ο συνήθως. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πολύ καλό και για τους άλλους. Κύριε Υπουργέ, ίσως ε, πρέπει να πω το εξής. Αυτά που είπατε είναι πολύ γνωστά. Θα ήθελα να ακούσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Τελικά, ποιος είναι πιο κοντά στην προσχώρηση, η Σοφία, η Σερβία ή το Μαυροβούνι ή η Μακεδονία. Ποιος είναι πιο κοντά στην ε, προσχώρηση. Ευχαριστούμε Υπουργέ. Ε, να σας και να σας πω ε, ποια χώρα εγώ θεωρώ ότι είναι πιο μπροστά από τις τρεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε στις διαπραγματεύσεις ούτε στην εκπλήρωση των κριτηρίων θα ισχύει αυτό και επίσης υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν διαφορετικές ταχύτητες μέχρι τελικά να ενταχθούν οι χώρες αυτές. Ευχαριστούμε Υπουργέ. Από ό,τι ξέρω πρέπει να φύγετε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λοιπόν λυπάμαι που πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν λόγω έλλειψη χρόνου ε, θα απαντηθούν γραπτά και ως εκ τούτου ολοκληρώνεται η ώρα των ερωτήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και κατόπιν τούτου λύεται η συνεδρίαση μέχρι τις 9 το βράδυ. Γεια σας.